Αγαπητοί συνάδελφοι, κάναμε το διάλειμμα μας. Ε, αναχώρησαν οι συνάδελφοι της Επιτροπής Περιβάλλοντος, οπότε θα συνεχίσω, θα δώσω δύο λεπτά στην εισηγήτρια, ώστε στο μεταξύ να κάνω τις ανακοινώσεις Μαρία, να προλάβετε να δείτε λίγο, να οργανωθείτε, διότι δεν έχουμε ακόμη κάνει τις ανακοινώσεις ε, για την Επιτροπή. Πρώτη ανακοίνωση την επόμενη Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου και θέλω βοηθεί και τα μέλη του προσωπικού να το σημειώσουν και να το στείλουν ε, στα μέλη. Στις 3 το μεσημερί θα έχουμε κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή ε, Εξωτερικών Υποθέσεων για να μιλήσουμε για την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών. Όπως γνωρίζετε η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται από πολλά ζητήματα, πρέπει να γίνουν εκλογές αλλά δεν γίνονται ε, ξέρουμε το θέμα με την αναστολή τη βοήθεια. Πολύ σημαντική λοιπόν η συζήτηση από κοινού με την ΑΦΕ την επόμενη εβδομάδα. Ελπίζω λοιπόν να έχουμε μεγάλη προσέλευση από του συναδέλφου. Και την επόμενη Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου, και εδώ παρακαλώ να ειδοποιήσετε τα μέλη από τις 12 μέχρι τη 1.30 στο χώρο Γεχοντι Μελουχίν η Επιτροπή ΔΕΒΕ θα φιλοξενήσει μαζί με την UNICEF και την DG ECO μια εκδήλωση για την εκστρατεία Emergency Lessons αφορά τα παιδιά που πλήττονται από τις επιπτώσεις των ε, ένοπλων συγκρούσεων. Θα έχετε δει όλοι τις εικόνες από το Χαλέπι στην τηλεόραση αυτό το Κυριακό. Τρομακτικές σκηνές, ε, καταστραμμένα νοσοκομεία, και πρέπει πραγματικά να επενέσουμε τους ανθρώπους της UNICEF που εργάζονται σε τόσο επικίνδυνες συνθήκες επί τόπου. Οπότε ελπίζω να προσέλθουν την επόμενη τρίτη οι συνάδελφοι ο, ο, από τις 12 μέχρι τη 1.30 ο Επίτροπος κύριος Στυλιανίδης θα βρίσκεται εκεί και ο Justin Forsyth, ε, αναπληρωτής εκτελεσμός διευθυντής της UNICEF και μετά στο Στρασβούργο. Έχουμε το βραβείο Σαχάροφ ε, κοινή συνέδριαση με την ΔΕΒΕ ΑΦΕΤ και ΝΤΡΟΑ ε, Δευτέρα το βράδυ στις 7 όπου θα απονεμηθεί το βραβείο Ζαχαρόφ στις ε, ε, για ζήτη που έψαν θύματα βία στη Συρία. Συνάντησα μία από αυτές τις νεαρές, πολύ νεαρές γυναίκες και πιστεύω ότι θα είναι εξαιρετικά συγκινητική η ιστορία που θα ακούσουμε από αυτές τις γυναίκες, ε, πόσο έχουν υποφέρει από αυτές τις τρομακτικές συνθήκες και όμως τις επιβίωσαν. Και ε, θα δούμε και πώς υποστηρίχθηκαν μετά για να ξαναφτιάξουν τις ζωές τους. Ε, Όλα τα μέλη γνωρίζουν από έτσι λοιπόν να... ποιες εκδηλώσεις έχουμε από τώρα μέχρι τα Χριστούγεννα. Να υπενθυμίσω ότι στις 5 σήμερα θα γίνει η κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Ελέγχου των προπολογισμών που θα λάβει η χώρα στην αίθουσα 1G2 και εκεί θα συζητηθεί θα συζητηθούν εκθέσεις από διάφορες αντιπροσωπείες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα διάφορα κράτη-μέλη για το πώς δαπανώνται ε, τα κονδύλια βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν επίμαχο το θέμα πέρυσι, οπότε τώρα κάνουμε μια συνάντηση για να δούμε ακριβώς τι γίνεται με την αναπτυξιακή βοήθεια. Ε, Όπω θα μαθαίνουμε από του πρέσβει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτέ είναι οι ανακοινώσει μου. Ε, τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρία δεν έχουμε δει ακόμα από το σημείο 3. Αν έχετε παρατηρήσει ε, ε, γνωστοποιήστε τα στη γραμματεία πριν το τέλο τη συνεδρία. Αλλιώ θα θεωρηθεί ότι εγκρίνονται. Στο σημείο 4, αποφάσει των συντονιστών, παρακαλώ δώστε οποιαδήποτε σχόλια στη γραμματεία, αλλιώ θα θεωρηθεί ότι έχουν εγκριθεί. Σημείο 25, ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα έρθει αύριο. Η Επιτροπή δεν ξέρω αν έχουμε άλλη ανακοίνωση από την Επιτροπή σήμερα. Όχι. Ωραία. Καμία λοιπόν. Αύριο θα έχουμε εδώ τον Επίτροπο. Οπότε μπορούμε να περάσουμε τώρα στο σημείο 7. Σημαντικό σημείο είναι η γνωμοδότησή μας ε, ε, που αφορά ε, για την Επιτροπή, Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την Ανιθαγένεια στην Νότια και Νοτιοανατολική Ασία, η συγκίτρια κυρία Μαρία Χόιμπουχ. Σημαντικό ζήτημα με το Ροχίνγκα και όλα τα ζητήματα αυτή τη στιγμή όσον αφορά την ανιθαγένεια, την τρομακτική φτώχεια και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στην περιοχή αυτή του Μιανμάρ και υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Λοιπόν, Μαρία, έχετε τον λόγο. Σε ευχαριστώ πολύ, Ελέντα. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρωτού σας ε, παρουσιάσω αυτή την έκθεση, θα ήθελα ε, να σας πω έτσι δύο λόγια ως προς το υπόβαθρο αυτής της ε, έκθεσης. Παγκοσμίω λοιπόν σήμερα υπάρχουν 10 εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι είναι ανιθαγενείς και ως ανιθαγενείς ορίζεται το πρόσωπο εκείνο το οποίο δεν αναγνωρίζεται από κάποιο κράτος με βάση τις νομοθεσίες του ως ε, επίκος. Και αυτό δηλαδή ορίζει και η σχετική σύμβαση των ΗΕ για τους ανιθαγενείς του 1954. Τώρα, το να γίνει κανείς ανιθαγενής μπορεί να οφείλεται σε διαφορετικούς ε, λόγους. Ε, και η έκθεση εδώ η δική μας στρέφεται προς πολύ συγκεκριμένες εθνοτικές πληθυσμιακές ομάδες ε, γιατί ε, εδώ βλέπουμε ε, συγκεκριμένα άτομα που ανήκουν δηλαδή σε μια θρησκευτική μειονότητα ή σε μια συγκεκριμένη εθνοτική μειονότητα ενδέχεται να αποκλειστούν από τη λήψη της ε, ηθαγένειας ενός κράτους. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι έχουμε ολόκληρες ομάδες ανθρώπων οι οποίες δεν καθίστανται ανηθαγένεις. Ένα παράδειγμα είναι οι Ροχίνια, οι οποίοι προέρχονται κατάγονται από τα δυτικά ε, της ε, Βερμανίας. Αλλά μετά από την σχετική ε, νομοθεσία που υιοθετήθηκε από την Βερμανία, το Μιανμάρ δηλαδή σήμερα του 1982 είναι πλέον επισήμως ανιθαγενείς και κατά συνέπεια αποτελούν τη μεγαλύτερη εθνοτική ομάδα ανιθαγενών σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι πραγματικά απίστευτο το ότι έχουμε δύο εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι δεν ανήκουν επισήμως σε κανένα κράτος. Δεν έχουν καμία ε, ηθαγένεια και το να μην έχει κανείς βέβαια επικότητα ενός κράτους έχει δραματικές επιστώσεις ε, στη ζωή του. Δηλαδή έχουν να αντιμετωπίσουν πολύ σημαντικές ε, δυσμενείς διακρίσεις στον τομέα της υγείας, της εκπαίδευσης και της εξέπρασης εργασίας. Ακόμα και η σύναψη ενός γάμου μπορεί να δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα. Άρα λοιπόν εκείνο που εγώ προσπαθώ να εξετάσω είναι ε, το τι μπορεί να γίνει σε επίπεδο αναπτυξιακής πολιτικής ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση των ανηθαγενών ειδικότερα δε στην ε, Νότια και Νότια-Ανατολική Ασία. Και προτείνουμε συγκεκριμένα. Όταν καταρχήν λύγεται Γίνεται λόγος για ανηθαγένεια και για τις καταστροφικές επιπτώσεις της ανιθαγένειας σε επίπεδο δηλαδή θεμελιωδών δικαιωμάτων, υποχρεώσεων ε, και δικαιωμάτων του πολίτη, ε, πρόσβαση σε περιουσιακά στοιχεία, πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες, ε, τότε θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η ανιθαγένεια έχει πολύ δυσμενείς επιπτώσεις για τις ε, προοπτικές ανάπτυξης των λόγω εθνοτικών ομάδων και κατά συνέπεια πολύ δυσμενείς ε, προοπτικές σε ό,τι αφορά και την ατζέντα του 2030. Η σχέση τώρα, και αυτό είναι ένα δεύτερο ζήτημα μεταξύ της ανεθαγένειας και των ε, κοινωνικών επιπτώσεων, δεν μπορεί να διαγραφεί ή να παραβλεφθεί. Κατά συνέπεια λοιπόν οι σχετικές κυβερνήσεις θα πρέπει να κληθούν να, να υιοθετήσουν μια δίκαιη νομοθεσία σε ό,τι αφορά τη χορήγηση ηθαγένειας ενώ θα πρέπει να προβλέψουν και ε, τις κατάλληλες δίκαιες και χωρίς διακρίσεις διαδικασίες για την καταχώρηση ε, των ε, κατοίκων τους. Ε, τρίτο στοιχείο που αναφέρουμε είναι ότι πρέπει να καλέσουμε τις κυβερνήσεις του Μπρουνέη, της ε, και άλλων να καταργήσουν την υφιστάμενη, τις υφιστάμενες διακρίσεις που ισχύουν στη σημερινή τους νομοθεσία. Για παράδειγμα, εάν οι γυναίκες δεν διαθέτουν το ίδιο δικαίωμα μεταβίβαση στις ηθαγένειές τους ε, στα παιδιά τους χωρίς καμία διάκριση ε, σε σύγκριση με τους άντρες. Θα πρέπει λοιπόν να καλέσουμε τις εν λόγω χώρες να βελτιώσουν σχετική νομοθεσία, να υπάρχει δηλαδή το δικαίωμα λήψης της ηθαγένειας ε, από τους γονείς τους των παιδιών. Ένα ακόμα στοιχείο είναι ότι θα πρέπει να τονίσουμε ακόμα περισσότερο την, ε, τη διάσταση του γεγονότος ότι ε, στις, ε, στην περίπτωση των περισσότερων Αθαγινών έχουμε να κάνουμε με πρόσφυγες ή εκδιωγμένους. Για παράδειγμα, 1,5 εκατομμύριο των ε, ανιθαγενών είναι ε, πρόσφυγες ή εκδιωγμένοι. Από εκεί και μετά ένα ακόμα σημείο είναι ότι θα πρέπει να επιτύχουμε ένα ενιαίο πλαίσιο ενιολογικό ορισμό, δηλαδή σε ό,τι αφορά την ανιθαγένεια. Σήμερα δεν υπάρχει ένα τέτοιο ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει κοινό ορισμό ε, για τον οποίο να δεσμευθούν όλες οι χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να, να συμπεριλάβει ω συστατικό στοιχείο τη αναπτυξιακή τη πολιτική ε, και στο πλαίσιο των συμφωνιών που συνάπτει σε επίπεδο εμπορική πολιτική τα ζητήματα τη ανηθαγένεια ε, σε ό,τι αφορά την περαιτέρω προώθηση τη ανάπτυξη, τη ειρήνη και τη σταθερότητα. Δεν ε, παρευρίσκονται βέβαια αυτή τη στιγμή πολλοί συνάδελφοι στην αλλά αν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα ήθελαν να σχολιάσουν, την έκθεση είναι πρόσδεκτα τα σχόλιά του. Ε, θεωρούμε πω είναι πραγματικά σημαντικό να δώσουμε φωνή σε αυτού του ανθρώπου, του αγενεί, ε, και να διασφαλίσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματά του ανά τον κόσμο. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Αν και δεν είναι πολλοί συνάδελφοι εδώ, θα ήθελα να πω ότι το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό. Οι Ροχιγκίγια είναι απάτριδες όχι μόνο στο Μιανμάρ, αλλά δεν τους επιτρέπεται να επιστρέψουν και στο Μπαγκλαντές. Όταν κανείς είναι άνηθα γεννήσει ή απάτρις, δεν έχει κράτος να, να επιστρέψει και να γυρίσει. Σαφέστατα υπάρχει καταστρατήγηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Έχουμε τον κύριο Χόρχε Τελασκαπελερία από τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης έχει δώσει πολιτική χρειά στο θέμα, έχει μιλήσει με τον Παγκλαντές ή τη Μιανμάρ. Και συμφωνώ και με τη Μαρία, πρέπει να ε, λυθεί, να αντιμετωπιστούν και τα ζητήματα απόλυτης φτώχεια για αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά ας ξεκινήσουμε την ε, γενική διεύθυνση, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αξιότιμη κυρία εισηγήτρια, αγαπητοί συνάδελφοι, με μεγάλη χαρά συμμετέχω εδώ σήμερα. Ξέρετε, η ανιθαγένεια επηρεάζει πάρα πολλούς ανθρώπους στην Νότια και Ανατολική Ασία. Η συγκήτρια αναφέρθηκε στον αριθμό των 10 εκατομμυρίων ανθρώπων. Έχει πάρα πολλές αιτίε, διακρίσεις μέσα στις εθνικές νομοθεσίες, ε, αυθαίρετη νόμη από οικειοκρατία. Ε, ξέρετε, η ιστορία της αποικιοκρατίας οδήγησε σε τέτοιου είδου φαινόμενα και τα παιδιά αυτό που έχουν υποστεί διακρίσεις έχουν υποστεί τις ίδιες. Η ανιθαγένεια εμποδίζει τους ανθρώπους να γίνουν καλύτεροι οι ίδιοι, να αποκτήσουν οντότητα, να αναπτυχθούν, να στηρίξουν την κοινωνία και να έχουν πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες όπως είναι η εκπαίδευση. Δεν μπορούν να δουλέψουν, να ταξιδέψουν και να έχουν πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Και μάλιστα ε, ε, για αυτούς τους λόγους παγιδεύονται ακόμα πιο εύκολα και ακόμα πιο γρήγορα στην παγίδα της φτώχειας. Όταν μιλούμε για ολόκληρες κοινότητες έχουμε δείκτες ανάπτυξης με καταστροφικές επιδόσεις και πολύ σημαντικές ανθρωπιστικές ανάγκες για ανθρωπιστική βοήθεια. Όπως και η συγγήτρια αναφέρει, είναι σαφέ αυτό το οποίο συμβαίνει στη Μιανμάρ. Η φτώχεια παραμένει στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μα. Ο κόσμος έχει αλλάξει όμως και υπάρχουν διάφοροι τρόποι να την αντιμετωπίσει κανείς. Έχουμε τη συνολική στρατηγική για την Ευρώπη και την ατζέντα για το 2030. Και καλό είναι να αναφέρω εδώ την πρόταση για μια νέα Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Ανάπτυξη κόσμος είναι πολύ πιο περίπλοκος, αντιμετωπίζει πιο πολλές προκλήσεις και είναι διασυνδεδεμένος. Οι μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη και η απάντηση που δώσαμε σε αυτές το δείχνουν αυτό και το αναδεικνύουν. Η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και η αντιμετώπιση των βασικών αιτιών μετανάστευσης είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Την περασμένη εβδομάδα οι δημοσίευσεις που έγιναν καλώς τονίζουν ότι Αποτελεί μέρος των αρχών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης η προσέγγιση μας για ε, την ανάπτυξη. Έχουμε εκεί το δικαίωμα μη διάκρισης, τη συμπερίληψη και τη συμμετοχή. Πάρα πολλά ε, άτομα που είναι απάτριδες τους αρνούμαστε, τους αρνούνται ε, τα δικαιώματα αυτά. Το σημαντικό είναι να μην μείνει κανείς πίσω και όλο αυτό θα παραμείνει στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής δράσης τα επόμενα χρόνια. Όμως, επειδή τα ζητήματα είναι τόσο περίπλοκα, για να αντιμετωπίσουμε την ανεθαγένεια πρέπει να έχουμε προσέγγιση πολυμερή και πολυσχεδή. Ανθρωπιστική βοήθεια και ενίσχυση της αναπτυξιακής συνεργασίας μπορεί να ελαφρύνει, να απαλύνει τις αρνητικές επιπτώσεις αυτής της κατάστασης. Ας είμαστε σαφείς όμως, χρειάζονται τέτοιου είδους παρεμβάσεις, είναι αναγκαίες και απαραίτητες, αλλά δεν εξαλείφουν τις αιτίες του κακού, το λόγο για το οποίο δημιουργείται η ανηθαγένεια. Θα ήθελα να αναφερθώ στα εργαλεία που αξιοποιούμε υπό αυτή την έννοια σήμερα. Τρία-τέσσερα σημεία εν συντομία. Πρώτον, με το Ευρωπαϊκό Εργαλείο, την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αυτό είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιούμε γιατί η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών είναι απαραίτητη για την χαρτογράφηση της κατάστασης και της βελτίωση της κατάστασης των Ροχίνγκια στις σχετικές αντίστοιχες χώρες. Ε, έγινε μια, μια προκήρυξη υποβολής προτάσεων για τη στήριξη των μεταναστών, των ετούντων άσυλο σε τρίτες χώρες, των εσωτερικώς εκτοπισμένων και των απάτριδων. Και αυτό αναφέρεται ρητός. Ως προς την ανιθαγένεια, στόχος είναι να προστατευτούν τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων να ε, ε, να υπάρξει επιχειρηματολογία επαρκής για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, να ε, υπάρξει διευθέτηση των φακέλων αυτών των ανθρώπων και να προληφθεί να μην υπάρξουν και άλλοι που να τους αποδοθεί αυτός ο χαρακτηρισμός. Αυτό είναι το εργαλείο της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε όμως και περιφερειακά προγράμματα, τα ξέρετε πολύ καλά. Το πρόγραμμα AUP Στηρίζουμε ε, υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και διαβίωσης ε, σε απάτριδες και θα θέλαμε να συμπεριλάβουμε αυτή τη διάσταση των ανιθαγενών κοινοτήτων στα περιφερειακά προγράμματα συνεργασίας που έχουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι πάντοτε εύκολο αυτό. Και υπάρχει διάκριση και υπάρχει ε, έλλειψη βούλησης από τη πλευράς πολιτικών αρχών και αυτό δυσκολεύει τις συζητήσεις. Υπ' αυτή την έννοια είναι σαφέστατη η ανάγκη οικοδόμησης διαλόγου. Για παράδειγμα, και είναι ένας από τους τρόπους που θα πρέπει να αξιοποιήσουμε ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Οι οικονομικές συμφωνίες και συμφωνίες χρηματοδότησης. Υπογράφουμε συμφωνίες χρηματοδότησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξεκάθαρα με αυτό το σκοπό. Θα πρέπει να τονίσουμε τη σημασία της εμάς τον πολιτικό διάλογο σε πολιτικό επίπεδο και για τη διαμόρφωση της πολιτικής με τις ε, από κοινού επιτροπές με τις εκάστοτε χώρες σε ό,τι αφορά το πόσο μαστίζεται η κοινότητα των ροϊνκά, είναι ένα ζήτημα υψηλής προτεραιότητας, το οποίο πράγματι τέθηκε και από την εισηγήτρια. Και αυτά ε, υπογραμμίζουν την ανάγκη για ε, δράση έτσι, στο πλαίσιο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Αξιοποιήσαμε λοιπόν αυτά τα εργαλεία για να απαλύνουμε τη μάστιγα που έχει πλέξει την κοινότητα αυτή των Ροχιγκίγια. Στηρίζουμε το πληθυσμό στη σχετική πολιτεία της Μιανμάρ και η Ευρωπαϊκή Ένωση άλλωστε είναι μία από τους βασικούς δωρητές στη χώρα αυτή. Δίνει ε, αναπτυξιακή βοήθεια ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι ασχολούμαστε και προσπαθούμε να εξαλείψουμε τις βασικές αιτίες ε, τις οποίες υφίσταται διακρίσεις και η βασική αιτία είναι η φτώχεια και προσπαθούμε να ελαφρύνουμε αυτό το καθεστώς της φτώχειας. Έχουμε συγχρηματοδοτούμενα τρία ε, ε καταπιστέματα για την ασφάλεια των τροφίμων, την επάρκεια, την ε, εκπαίδευση και την υγεία και δίνουμε βοήθεια στην πολιτεία στο κρατήριο του Ρακάν. Στο, στη βόρεια περιοχή του Ρακάν, όπου διαβεί και η μεγάλη πλειοψηφία αυτού του πληθυσμού, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί ένα project 15 εκατομμυρίων ευρώ. Care και Action contre la faim σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες. Έχουμε δώσει εκπαιδευτική συνδρομή μέσω μιας χρηματοδότησης διμερούς ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ ε, που απευθύνεται το πρόγραμμα αυτό στα παιδιά που διαβιούν στο Βορρά. Βλέπετε λοιπόν πώς παρεμβαίνουμε, παρεμβαίνουμε αξιοποιώντας όλες μας τις δυνατότητες σε αυτό το συγκεκριμένο γεωγραφικά τόπο που διαβεί η συγκεκριμένη κοινότητα ανθρώπων. Θα ήθελα να επιμείνω για άλλη μια φορά στο γεγονό ότι αυτό είναι μόνο ένα από του τρόπου αντιμετώπιση του προβλήματο. Όπω ανέφερα και προηγουμένω, είναι αδύρυτη σημασία, είναι πολύ μεγάλη σημασία ο πολιτικό διάλογο και γι' αυτό έχουμε ε, προτάσει ψηφισμάτων για τη Μιανμάρ ε, και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και σε επίπεδο Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Εθνών. Ε, ε, υπάρχουν τακτικές επισκέψεις στο κρατήδιο του Ρακάν έτσι ώστε να παραμείνει το θέμα ψηλά στον κατάλογο προτεραιοτήτων κατά τις διαβουλεύσεις και τις συνομιλίες με όλες τις σχετικές αρμόδιες αρχές. Της 22 Νοεμβρίου με την ευκαιρία της ε, τρίτης συνεδρίασης υψηλού επίπεδου Ευρωπαϊκής Ένωσης Μιανμάρ για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, εθίγει πάλι το ζήτημα. Αυτή ήταν και η πιο πρόσφατη παρέμβαση. Βεβαίω, υπάρχουν και άλλε χώρε, και θα ήθελα εν συντομία να αναφερθώ στον Παγκλαντέ, στο Νεπάλ και την Ταϊλάνδη. Στον Παγκλαντέ δίνουμε στήριξη στον πληθυσμό για στα στρατόπεδα, στου καταβλισμού των προφύγων για τη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσή του. Δουλεύουμε με την ε, υπάτη των ΗΕ για του πρόσφυγε, 20 εκατομμύρια ευρώ είναι ο χρηματοδοτικό φάκελο για την παροχή προστασία, ασφάλεια, βασικών υπηρεσιών και Στόχος είναι να στηρίξουμε εκεί 32.000 πρόσφυγες που ανήκουν σε αυτή την πληθυσμιακή κοινότητα. Έρχομαι τώρα στο Νεπάλ και να πω ότι για πάνω από δύο δεκαετίες παρεμβαίνουμε στο Νεπάλ. Είναι με μεγάλη η ιστορία και στηρίζουμε πρόσφυγες από τον Μπουτάν. Ε, αρχικά 120.000 πρόσφυγες ζούσαν εκεί και έχουμε καταφέρει μετά από δύο δεκαετίες να έχουμε μόνο 13.000 πρόσφυγες από το ε, Πουτά να συνεχίσουν να διαβιούν στους καταπλησμούς των προσφύγων. Ε, είναι πολύ μικρό το νούμερο αυτό και συνέχισε η δουλειά, η εργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό σε συνεργασία με την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία των ΗΠΑ για τους πρόσφυγες. Τα νούμερα βεβαίω είναι μικρότερα, αλλά παραμένει σημαντική η παρουσία των προσφύγων από το Μπουτάν για την προστασία των δικαιωμάτων τους, για την ασφάλειά τους, για την κάλυψη των βασικών τους αναγκών. Δεν έχουν λησμονηθεί. Και τέλος για την Ταϊλάνδη, την οποία αναφέρει, ε, ε, η οποία αναφέρεται στην εισήγηση, έχουμε ε, συστήσει και δημιουργήσει ένα πρόγραμμα ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ που ασχολείται με θέματα διαβίωσης, εκπαίδευσης, υγιεινής, υγείας. Ε, ε, ε, δικαιούχοι είναι πρόσφυγες που μένουν σε νέα καταβλισμούς στα σύνορα και τις γύρω κοινότητες, την τοπική κοινότητα. Πράγματι η Ροχινγκία είναι περίθωροποιημένη στη Μιανμάρ και οι μουσουλμάνοι αποτελούν εν γέννη στόχο. Επομένως στόχος μας είναι η στήριξη των ευπαθών πληθυσμών. Σε κάθε περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση σε πάρα πολλά μέρη έχει προσφέρει στήριξη. Θα μπορούσα να αναφερθώ ακόμα και στη μειονότητα των Χμέρ στο Βιετνάμ και την προσπάθεια αυτών να αποκτήσουν βιετναμέζικη υπηκότητα και να βελτιώσουν τις συνθήκε ζωή του. Σε κάθε περίπτωση το σημαντικό και ελπίζω να συμφωνήσετε είναι να στηρίξουμε τους ανθρώπους όχι μόνο από την ηλική σκοπιά ή την οικονομική σκοπιά, αυτό το κάνουμε με τα διάφορα προγράμματα και σχέδιά μας, αλλά ε, να υπάρξει και πολιτική δέσμευση, πολιτική βούληση και εκστρατεία ευαισθητοποίησης. Η Επιτροπή συνεχίζει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να είναι παρούσα σε πολλά μέρη στον κόσμο για να αντιμετωπιστεί το θέμα των απάτριδων. Ε, το επιδιώκουμε αυτό και το επιτυχάνουμε μέσα από τα περιφερειακά μας προγράμματα τα οποία έχω αναφέρει επανειλημμένως και άλλωστε είναι πρόθεσή μας αυτή το σκέλος, αυτή τη διάσταση να τη περιλαμβάνουμε όλο και περισσότερο στις τακτικές και συνηθισμένες δραστηριότητες συνεργασία σε θέματα αναπτυξιακά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχει κάποιος κάτι να προσθέσει. Ναι, αν με επιτρέπετε κυρία Πρόεδρε να προσθέσω κάποια πράγματα για την κατάσταση των Ροχέγγια και το, για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, για το θέμα αυτό. Όπως είπε μόλις ο συναδέλφος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση ε, κάνει συνεχίσει εκκλήσεις στην κυβέρνηση του Μιανμάρ να αντιμετωπίσει τις αιτίες της κατάστασης ε, στην περιοχή Ρακάν και αυτό έχει αναφερθεί σε πολλά συμπεράσματα του Συμβουλίου ε, για το Μιανμάρ από το 2013 σε μια πρόσφατη κοινή ανακοίνωση για τη Μιανμάρ είπε ότι εκπρόσωπος ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσαν μια κοινή ανακοίνωση 1η Ιουνίου όπου έθεσαν τα ανθρώπινα δικαιώματα ως ε, βασικό ε, σημείο δέσμευσης μαζί με το Μιανμάρ και στο πλαίσιο των προτινόμενων πρωτοβουλειών ζητάμε εξάλληψη της ε, ανηθαγένειας και ίσα δικαιώματα για όλους τους πολίτες καθώς και έκδοση εγγράφων ταυτότητας. Και αυτό το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό διότι αυτή τη στιγμή ένα σημαντικό πρόβλημα στο Μιανμάρ είναι η έλλειψη παντός είδους εγγράφου για τον ανιθαγενή πληθυσμό των Ροχίνγκια. Δεν γίνεται καν καταγραφή ε, των ανθρώπων. Αυτό που βλέπουμε ουσιαστικά είναι μια παρατεταμένη ανθρωπιστική κρίση με ρίζες ε, σε ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στα πιο πρόσφατα συμπεράσματα του Συμβουλίου για το Μιανμάρ γίνεται έκκληση για μια ευρωπαϊκή στρατηγική όσον αφορά τη Βερμανία, το Μιανμάρ. Στις 22 Ιουνίου φέτος και εκεί αναφέραμε το ζήτημα αυτό. Εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σημειώνει ικανοποιητικά τις προσπάθειες του Μιανμάρ ε, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων ε, και τις καταστάσεις των Ροχίνγκια. Αυτό συμπεριλαμβάνει πολιτικές διαδικασίες ε, με την επίλυση της ανιθαγένειας πολλών ατόμων με μη διακριτικό τρόπο μέσω μιας διαφανούς ε, διαδικασίας ε, δίνοντας τέλος στον εκτοπισμό. Αυτό είναι το βασικό θέμα στο οποίο εστιαστήκε και η επίσκεψη μας πέρυσι στο Μιανμάρ κατά την οποία διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Ένωση τον ανθρωπιστικό διάλογο με επικεφαλής της αντιπροσωπείας τον κύριο Σταύρο Λαμπρινίδη και δεδομένων των τελευταίων εξελίξεων της έντασης της βίας στην περιοχή το θέμα δεν ήταν μόνο διαλογός για τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και διμερείς συναντήσεις με πολιτικούς παράγοντες της χώρας. Εδώ ο ειδικό εκπρόσωπο συναντήθηκε με του ε, ε, ομολόγους του και έστειλε ηχηρό μήνυμα ότι εκτός από την αντιμετώπιση των εκτέκτων αναγκών, ε, των επικουσών αναγκών του πληθυσμού Ροχίνγκια, οι υπό τις συνθήκες, είναι επίσης πολύ σημαντικό η κυβέρνηση να συνεχίσει με το να καθορίσει τις πολιτικές προτεραιότητες που είχε ξεκινήσει από τότε που ανέλαβε καθήκοντα τον Απρίλιο φέτος. Τότε είχαμε δει ήδη κάποιες πολιτικέ ε, ε, πολιτικές ανακοινώσεις από την Άουνγκ Σανσούτσι, τη δημιουργία μιας κεντρικής επιτροπής ε, για ένα διπουργικό οργανισμό ο οποίος θα επιδίκει να βρει μια βιώσιμη λύση Ήδη έχει εκδώσει 142 συστάσεις αυτό ο διακυβερνητικός οργανισμός για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Αλλά το πιο ενθαρρυντικό ήταν η δημιουργία, ήταν μια συμβουλευτική επιτροπής με τον Κόφι Ανάν ε, ως ε, πρόεδρο και άλλα δύο ε, ξένα μελή και επτά μέλη από τη Μιανμάρ με ε, καθήκον αυτής της Επιτροπής το να βρει βραχή πρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ε, ε, λύσεις για τα δεινά του πληθυσμού αυτού στην πολιτεία Αρακάν. Αλλά η κυβέρνηση αυτή ξεκίνησε μια διαδικασία επαλήθευσης ηθαγένειας τον Ιούνιο. Ωστόσο η διαδικασία αυτή δεν έφερε αποτελέσματα λόγω τη ε, έλλειψης πληροφοριών αλλά και εμπιστοσύνη ε, τοπικά. Οπότε οι ΗΠΑ ε, ενθάρρυναν την κυβέρνηση τη Μιανμάρ στι διάφορες συναντήσεις να ξεκινήσει μια ενημερωτική εκστρατεία ώστε να βελτιωθεί η εμπιστοσύνη και από τον πληθυσμό Ροχίνγκα στα λόγω αναμένουμε λοιπόν να δούμε τι αποτέλεσματα θα έχουν όλα αυτά στο μέλλον. Αλλά όπως ανέφερα, το μήνυμα ήταν σαφές ότι για την περιοχή Αρακάν να από την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τις βασικές αιτίες, τις ρίζες της κατάστασης. Ευχαριστούμε. Είναι θετικό το γεγονός ότι λαμβάνονται τόσες δράσεις γιατί ίσως ε, κάποτε να μην έχουμε τόσες ε, συγκρούσεις. Ε, Ίσως δηλαδή να δώσουμε κάποια προοπτική σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ξέρω κατά πόσο, Μαρία, θες να σχολιάσεις. γιατί κάπου εκεί στη, στο σχέδιο ψηφίσματο γίνεται μια αναφορά στα όσα σχέδια τα οποία έχει θέσει εκείνη η Επιτροπή. Οπότε ενδεχομένω θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε κάτι, κάτι σχέση με αυτό. Λόγω σε εσένα, Μαρία. Σε ευχαριστώ θερμά, Λίντα, και ευχαριστούμε και του εκπροσώπου τη Επιτροπή για όλε τι ενημερώσει. Ε, χαιρετίζομαι κάθε είδου ε, περαιτέρω πληροφορίε ε, τόσο για του Ροχέγγα όσο και για όλου του υπολείπου ανθρώπου οι οποίοι ζουν σε αυτό το αβέβαιο καθεστώ του απάτριδα ή το ενθαγενή. Ε, προφανώς πρόκειται για ένα περίπλοκο πρόβλημα για το οποίο δεν υπάρχουν εύκολε λύσει, αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε ότι πραγματικά ε, πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο ε, ε δεν βρίσκεται έτσι, δεν τραβάει τα φώτα, φώτα της δημοσιότητας και το ξεχνάει η κοινή γνώμη. Εμεί, λοιπόν είμαστε ένα ε, κοινοβούλιο και κατά συνέπεια θα πρέπει να μα απασχολήσει ένα τόσο σημαντικό θεμελιώδη ζήτημα όπως τις Ε, Πραγματικά θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε δώσουμε και πάλι λίγη ορατότητα σε αυτό το ζήτημα μέσω και ενό νέου ψηφίματο για να δώσουμε και ε, φωνή σε αυτού του ανθρώπου. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια καλή νομοδότηση από την πλευρά μα ε, και αναμένω με ενδιαφέρον τι ε, προτάσει των συναδέλφων. Και πραγματικά ελπίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε προ το καλύτερο τη ζωή αυτών των ανθρώπων. Ευχαριστούμε την Μαρία Χόιμπο και την Επιτροπή η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 7 Δεκεμβρίου, 7 Δεκεμβρίου το μεσημέρι. Καλώς λοιπόν κλείνουμε αυτό το τμήμα της συνεδρίασής μας εδώ σε αυτή την αίθουσα και θα συνεχίσουμε αύριο στις 9 το πρωί για να, να μεταφερθούμε στην αίθουσα ESP 1G2, 2 δηλαδή ορόφους ε, πιο κάτω όπου έχουμε την κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού στι 5. Ε, Κάποιους λοιπόν θα σα δω εκεί, του υπόλοιπου αύριο στι 9 το πρωί. Ευχαριστώ και του διερμηνείς.